versuchen wir Πολύ ωραία. Πολύ Ας το ξαναπροσπαθήσουμε λοιπόν, γιατί από ό,τι μου ανακοινώνουν μα ε, ακούνε πλέον και οι διερμηνεί. επιβεβαιώνουμε. Έχετε λοιπόν διερμηνία, κύριε και κύριοι, φανταστικά, πάρα πολύ ωραία. Κυρίε και κύριοι, α ξεκινήσουμε λοιπόν. Στις 9 Μαΐου, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η μέρα της Ευρώπης. Ο Ρόμπερτ Σούμαν με την ε, περίφημη διακήρυξη του ε, Σούμαν έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και εξ όσων γνωρίζω, τότε δεν υπήρχε η σύνδεση με την ημέρα αυτή, αλλά Σήμερα συνεδριάζει το Κοινοβούλιο στην, ε, στο Στρασβούργο και γι' αυτό λοιπόν σας καλωσορίζω και σε αυτή την εορταστική συνεδρίαση, σε αυτή την ημέρα της ε, Ευρώπης, την ημέρα Σούμαν. Μία ημέρα κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον Άνθρακ και το Χάλιβα έθεσε τις ε, αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τεχνολογικής άποψης, αλλά Έχουμε και το τεχνολογικό ζήτημα, αλλά θα ακούσουμε καταρχά ε, του κυρίε και κύριοι από την ε, Ορχήστρα του που Θα μα κάνουν μια μικρή μουσική εισαγωγή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι από το Οδείο του Στρασβούργου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έξοχη αυτή εισαγωγή. Αξιότιμοι συνάδελφοι, στις ε, ε, 9 Μαΐου του 1950, ο Ρόμπερτ Σούμαν είπε τις δύο αυτές τις φράσεις. Η διεθνής ειρήνη δεν θα μπορέσει να διατηρηθεί χωρίς ε, προσπάθειες ε, αντίστοιχες της απειλής που μας, ε, που με την οποία μας αντιμετωπεί η Ευρώπη δεν θα οικοδομηθεί με μιας. Και θέλει επίσης και συγκεκριμένες πράξεις για να μην υπάρξει η αλληλεγγύη στην πράξη. Σήμερα λοιπόν η Ευρώπη περνάει από μεγάλες τρικυμίες και ίσως να είναι και εν ώψη μιας ε, αποφασιστικής ε, στιγμής ρήψης και πιο πολύ από ποτέ το θάρρος ε, των πολιτών οι οποίοι δεσμεύονται για την Ευρωπαϊκή Ενότητα χρειάζεται και θα πρέπει να μας υπενθυμίσει το ότι είναι πραγματικά σημαντικό. Κάποια από τα πράγματα λοιπόν αυτά θα ήθελα να σας τα αναφέρω, να σας τα παραθέσω που μας υπενθυμίζουν κάποιοι ότι είναι πραγματικά σημαντικό η ειρήνη, η αλληλεγγύη και ο αμοιβαίος σεβασμός, ο αλληλοσεβασμός. Είναι σημαντικά λοιπόν τα τρία αυτά στοιχεία της ειρήνης, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. Θα πρέπει να τα εμβαθύνουμε να τα εμβαθύνουμε και να εμβαθύνουμε όχι σε αυτά που μας χωρίζουν, αλλά να εμβαθύνουμε σε αυτά που μας ενώνουν. Κυρίε και κύριοι, είναι... έχει αυτή στιγμή να αγωνιστούμε για την Ευρώπη αυτή. Δεν ε, μπορούμε να μας αφήνουν να, αφήνουμε να μας οδηγούν οι εχθροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται θάρρος και τόλμη και με θάρρος και τόλμη θα πρέπει να προχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Την προηγούμενη Παρασκευή είχα την ευκαιρία στο Βατικανό να ακούσω τον ε, Παπαφρακίσκο όταν έθεσε το ερώτημα του τι έγινε με την Ευρώπη, τι έχει συμβεί με την Ευρώπη, τι έχει συμβεί με την Ευρώπη του ουμανισμού, την πρωταθλήτρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τι έγινε με την Ευρώπη σας λοιπόν, με ρώτησε ο Πάπας με την πατρίδα των ποιητών, των φιλοσόφων, των μουσικών, των ε, ανδρών και γυναικών της επιστήμης. Τι έχει συμβεί λοιπόν με την Ευρώπη, τι συνέβη με την Ευρώπη των λαών και των εθνών, των μεγάλων ανδρών και γυναικών που είχαν το θάρρος και την τόλμη να ορθώσουν τον ανάστημά τους και ήταν μάλιστα αντιτεθειμένοι ακόμα και τη ζωή τους την ίδια να θυσιάσουν για την αξιοπρέπεια των αδελφών τους για να προασπιστούν αυτή την αξιοπρέπεια. Ο Πάπας λοιπόν μας είπε ότι θα πρέπει να στραφούμε και πάλι στους προπάτορες της Ευρώπης, αυτούς που ίδρυσαν την Ευρώπη. Γιατί αυτοί ήταν πρόθυμοι, ήταν τεθειμένοι να βρουν εναλλακτικέ νέους τρόπους να βρουν για να προχωρήσουν σε ένα κόσμο ο οποίος ε, είχε περάσει τη φρίκη του πολέμου των πολέμων. Και αυτό όχι επειδή είχαν μία ιδέα μόνο για την Ευρώπη, αλλά γιατί τόλμησαν, τόλμησαν να καινοτομήσουν, να φέρουν ένα νέο μοντέλο, ένα νέο μοντέλο για την ειρήνη και τη συνεργασία. Για να αντικαταστήσουν, να αντικαταστήσουν το μοντέλο της βίας και της φρίκης, στο οποίο είχαν ζήσει, στο οποίο είχαν μεγαλώσει. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή για να αγωνιστούμε για την Ευρώπη αυτή. Δεν πρέπει να αφήσουμε να ηγηθούν και να μας παραπλανούν οι πολέμοι της Ευρώπης. Μπορούμε και πρέπει με θάρρος και τόλμη και φιλοδοξία να συνεχίσουμε να προχωράμε την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Στις 26 Νοεμβρίου του 2014 ένας μεγάλος άνδρας, Dr. Τένις βρέθηκε εδώ στο κοινοβουλίο μας και είπε το εξής. Σε έναν κόσμο όπου αντιστρέφονται οι αξίες, όπου η βία είναι κάτι το καθημερινό και το συνηθισμένο, που παίρνει μορφές η βία που δεν θεωρούσαμε ποτέ ότι θα ήταν δυνατόν, θα πρέπει να αρθώσουμε τον αστυμά μας και να αντισταθούμε. Και θα πρέπει σε αυτόν τον δρόμο να κινηθούμε. Ο Δόκτωρ Μουκβέντε, μας είπε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν από μόνα τους τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Αποτελούν και ένα αντικείμενο που μας προκαλεί θάρρος και μας δίνει τόλμη και θα έπρεπε να σας δίνει τόλμη και εσάς στις εξωτερικές σας σχέσεις. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τα θεωρείτε ένα εργαλείο, ένα μέσο για την ανάπτυξη και την ειρήνη και σε άλλα μέρη του κόσμου για την δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε άλλα μέρη του κόσμου. Και εκεί λοιπόν, εδώ μάλλον στην αίθουσά μας αυτή, στο μικυκλίο μας, αυτός ο μεγάλος γιατρός, ο οποίος και τιμήθηκε και με το βραβείο Ζαχάροφ μας υπενθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί για αυτόν την ελπίδα. Την ελπίδα προκειμένου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα να έλθουν και στην δική του χώρα. Και είναι πιο σημαντικά αυτά από οποιαδήποτε οικονομική και χρηματοοικονομική ανησυχία και στις 3 Φεβρουαρίου του 2016 ο Νιγηριανός πρόεδρος Μπουχάρη εδώ πάλι μας δήλωσε ότι τα προβλήματα τα δικά σας είναι η κατανομή του πλούτου. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Το δικό μας το πρόβλημα όμως είναι η φτώχεια. Οι αρρώστιες και η υποανάπτυξη από τεχνολογικής άποψης. Γιατί τα ξεχνάμε αυτά τα λόγια τόσο γρήγορα. Όλα αυτά τα οποία επιδιώκουν για τους λαούς τους αυτοί οι άνδρες ή για τους ασθενείς τους, εμείς τα έχουμε κάθε μέρα, είναι αυτονόητα για μας. Και γι' αυτό λοιπόν έχει έρθει η στιγμή να πολεμήσουμε για την Ευρώπη. Δεν πρέπει να μας τρομάζουν οι πολέμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει με φιλοδοξία να προαγάγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πορτογάλος Πρόεδρος στις 12 Απριλίου δήλωσε το εξή και μιλώ στα πορτογαλικά. Είπε λοιπόν ότι ανήκει σε, ανήκω σε μια γενιά ο, για την οποία η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα όνειρο για την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρώπη την οποία ονειρεύομαι. Η Ευρώπη λέγω την οποία ονειρεύομαι, αυτή η οποία τόσες φορές έχει θριαμβεύσει υπέρ του, του και της βαρβαρότητας, θα ξεπεράσει και το θρησκευτικό φανατισμό και την τρομοκρατία. Ο άντρας λοιπόν αυτός, ένας ε, υπέρμαχος ένθερμος της ευρωπαϊκής ε, ολοκληρωσής, που είπε αυτά τα λόγια εδώ στο ημικύκλιο εξελέγησε στον πρώτο γύρο με συντριπτική πλειοψηφία στη χώρα του ως πρόεδρος. Αυτό τι καταδεικνύει ότι η δημοκρατία δεν σημαίνει να είναι κανείς κατά της Ευρώπης, αλλά μπορεί κανείς και υπέρ της Ευρώπης να υποστηρίζει την Ευρώπη και να εκλεγεί. Και κυρίες και κύριοι, έχει έρθει η ώρα πραγματικά να πολεμήσουμε για την Ευρώπη. Ο Τόμας Ήλβες, ο πρόεδρος της Εστονίας, στις 2 Φεβρουαρίου μας απέφθινε το λόγο και δήλωσε ότι είτε είναι η μετανάστευση, η μετανάστευση είτε είναι το ευρώ, είτε και οι στρατιωτικές επιθέσεις ε, για να μην μιλήσουμε για την απειλή της, τεχνο, της τεχνολογικής αλλαγής οι λύσεις που θα μας, θα μας επαναφέρουν σε, στα έθνη κράτη θα μας ε, πάνε πίσω στο χρόνο, σε μια εποχή όπου η έλλειψη φιλοδοξίας ε, θα οδηγήσει σε απώλεια για όλους, δίχως αμφιβολία. Θα επιστρέψουμε σε μια εποχή όπου θα επικρατήσουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Μια εποχή την οποία έχουμε δει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές ε, στην ιστορία. Και μιλάμε για τον πρόεδρο μιας χώρας ε, που γνώρισε την κομμουνιστική δικατορία και κατάφερε να την νικήσει με την εξέγερση των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ένταξε τη χώρα αυτή και έδωσε σταθερότητα, ασφάλεια και ειρήνη και κατάφερε λοιπόν ο πρόεδρος της Εστονίας να τα εξασφαλίσει αυτά για το κράτος τους. Η επάνωδος λοιπόν στα κράτη-έθνη μας ε, λέει ο πρόεδρος αυτός της μικρής αυτής χώρας η αναφορά σε μια τέτοια ανοτροπία θα μας ξαναφέρει στην εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από πλευράς ανοτροπίας και εγώ πιστεύω λοιπόν ότι έχει δίκιο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πολεμήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση αυτή την ημέρα Σούμαν. Μια ημέρα που δεν υποστηρίζεται αυτόματα το ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά είμαι πεπισμένο απόλυτα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στην Ευρώπη εξακολουθεί να υποστηρίζει την συνεργασία των εθνών και των κρατών πέρα από τα σύνορα με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε μια εποχή όπου βιώνουμε μια κρίση αλληλεγγύης όπου η κοινή βάση αξιών μας κλειδονίζεται τέτοιες εποχές λοιπόν θα πρέπει να θυμόμαστε την έκκληση τέτοιων ανδρών και γυναικών, την έκκληση του Ρόμπερτ Σούμαν ότι θα οικοδομηθεί η Ευρώπη σε μία ημέρα και ότι ε, στηρίζεται στην αλληλεγγύη στην πράξη. Όλα αυτά θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε κυρίε και κύριοι. Έχει έρθει η στιγμή να αγωνιστούμε για την Ευρώπη. Όλοι, όλοι, όλες οι Ευρωπαίε, όλοι οι Ευρωπαίοι. Γιατί το μοντέλο αυτό τη ε, διεθνικής δημοκρατίας έχει αποτεχθεί το καλύτερο μοντέλο για την εξασφάλιση τη Ειρηνή και τη ασφάλεια. Και όποιοι το πιστεύουν αυτό, του καλώ να σηκωθούν και να μην ε, σιωπούν πλέον και να δηλώσουν την υποστήριξή τους προς την Ευρώπη μας ανοιχτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Τα πρακτικά της 26ης ε, και 27ης